μια ευκαιρία στο Πακιστάν μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων καθώς ε, νομίζω πως ε, βρίσκεται σε καλό δρόμο και μάλλον θα υπογράψει και τη συνθήκη της Γενέβης. Σας ευχαριστώ. Περαιούτη η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Καζάκ για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Καλωσορίζω τον Επίτροπο κ. Ντεχούχτα και ευχαριστώ την κυρία Μάλστρομ. And as we are used, Καταρχάς δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Καζάκ. Τέσσερα λεπτά κύριε Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος λόγος ε, της έκθεσης είναι ότι η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους της Ένωσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, πρόκειται για την 17η οικονομία στον κόσμο, την έκτη στην Ευρώπη και τον 7ο εταίρο της Ένωσης σε εμπορικά ζητήματα. Οι ανταλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έφτασαν το 2008 στο το στο υψηλότερο όριο με 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, η έκθεση τονίζει τα εξής συνοπτικά. Πρώτον, παρά την Τελωνιακή Ένωση του 86 που επετέλεσε μεγάλη επιτυχία για την, για την ενοποίηση της, ε, των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχουν ακόμα μη δασμολογικά εμπόδια που πρέπει να υπερβεί η Τουρκία το συντομότερο δυνατό. Δεύτερον, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις ε, δεσμεύσεις της έναντι της Τουρκίας στον τομέα του εμπορίου και να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την πλατφόρμα της Μεκτής Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Μεκτής Επιτροπής Τελωνιακής Ένωσης. Η Τουρκία από την πλευρά της πρέπει να θέσει πέρα στις διακριτικές συμπεριφορές με ένα πλονέκτημα 15% για τους Τούρκους ανάδοχους στις δημόσιες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες με τις οποίες η Τουρκία δεν έχει ακόμα συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Πρόκειται για ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζει η Τουρκία για να συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να εξασφαλίσουν την ένταξη της Τουρκίας, ε, στη, τη συμπερίληψη δηλαδή της Τουρκίας, σε μελέτες ε, αντικτύπου τέτοιων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Επίσης, η παραποίηση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στις διμερείς ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο την διεθνή νομο και εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό, ιδίως σε ζητήματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Έκτον, θα έλεγα ότι η Τουρκία είναι μια πολύ ε, μια περιφερειακή δύναμη με μεγάλη επίδραση στην Μαύρη Θάλασσα και στον Κάφκασο. Νέες αγορές με πολλές δυνατότητες που θα συνέβαλαν στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ένωσης και της περιοχής αυτής. Τρίτον, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι δραστηριότητε των γυναικών σε παράλληλε δραστηριότητε. Αυτό το αποτελεί μια πρόκληση για την Τουρκία, η οποία οφείλει να λάβει σχετικά μέτρα. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες θεωρήσεων, χορήγησης θεωρήσεων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επιχειρηματιών και οδηγών φορτηγών από την Τουρκία. Η Επιτροπή δε πρέπει να παρακολουθεί κατά πόσο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά. Επιτρέψτε μου να, μάλλον ελπίζω να δεχθείτε ότι δύο τροπολογίες που υπέβαλα στατιστικού χαρακτήρα και ένα σύντομο σχόλιο για το πρόσφατο δημοψήφισμα και την επερχόμενη συνταγματική ε, αναθεώρηση που θα ολοκληρώσει την, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ελπίζω αγαπητοί συνάδελφοι η συζήτηση να αντικατοπτρίσει το πνεύμα συνεργασίας και το επικοδομητικό πνεύμα που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτές, να ευχαριστήσω τον κύριο Καζάκ διότι συνέταξε αυτή την τόσο ολοκληρωμένη έκθεση όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Επίσης να ε, συγχαρώ και τα μέλη τη Κοινοβουλευτική επιτροπή γιατί συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με την Ελληνική Ένωση ε, και τα άλλα θέματα επίση καλύπτονται όπω οι θεωρίε διαβατηρίων, οι, οι οδικές μεταφορές που δεν με αφορούν άμυνα στο χαρτοφυλακιό μου. Πρόκειται για κάποια πάρα πολύ σημαντική χώρα, σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο έβδομο εμπορικό εταίρο τη Ένωση και εμεί είμαστε επίση σημαντικό εταίρο για την Τουρκία. Ε, Έχουμε την Ελληνική Ένωση, έχουμε σημαντικές εμπορικές αλλαγές και είναι βέβαια και υποψήφια χώρα. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους πρόκειται για μια μοναδική ξεχωριστή σχέση. Τώρα έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τις εμπορικές σχέσεις, το οποίο είναι αυτή η Τελωνική Ένωση. Ακριβώς όπως λέει και η έκθεση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ένωση, ούτως ώστε να αναπτυχθεί το διμερές εμπόριο και να ωφεληθούν και τα δύο μέρη. Όμως, ή ακόμη εκκρεμούν κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα, διότι δεν έχει μπορέσει Τουρκία ακόμα πλήρως να εφαρμόσει τα τάους επιτάσεις στην Ελληνική Ένωση, οπότε δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, τα οποία κρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση 100% ε, ετήρησε τα όσα λέει η Ελληνική Ένωση από τη δική της πλευρά και οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συνολικές συμφωνίες που θα καλύψουν κάποια θέματα υπηρεσιών, κάποιους δημόσιους διαγωνισμούς ε, αλλά οι προτάσει μα δεν είναι αποδεκτέ από την ε, Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει τα διεύματα που χρειάζεται τόσο ώστε να ξεσορροπήσουν σχέσεις μας στον εμπόριο με την Τουρκία, όλα θα πρέπει και η Τουρκία να προχωρήσει όσον αφορά τι συμφωνίε ελευθερών εμπορίου με τι τρίτε χώρε και θα πρέπει να συνηθούμε με τους Τούρκους εταίρους όσον αφορά αυτές τις δημοτεύσει στις τρίτες χώρες. Και θα πρέπει να γίνουν και οι μελέτε των ε, επιπτώσεων για αυτές τις συμφωνίες. Εμείς σε τακτά διαστήματα προσπαθούμε να εξωθήσουμε την Τουρκία να, προ... επιλύσει αυτά τα προβλήματα και επίσης ε, όσον αφορά αυτούς που έχουν ε, συμφωνίες ελευθερών εμπορίου προς τα εκεί να προχωρήσουμε γιατί θέλουμε η συμμετοχή της Τουρκίας εκεί να γίνεται με κάποια προσερτημένη δήλωση ή με κάποιο άρθρο στο σώμα της συμφωνίας. Όμως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και αυτό είναι φιλιβάρο το οποίο ισχύει πλέον τη Τουρκία, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να υπάρχει εύρεθμη λειτουργία σε αυτή την Τελωνική Ένωση, Ένωση Τουρκίας. Επίση, θα πρέπει να σα πω ξεκάθαρα ότι υπάρχουν κάποιε αντιστάσει, κάποια προθυμία του Τουρκία, ώστε να εφαρμόσει πλήρως την Τελωνική Ένωση και αυτά όλα τα λέει η έκθεση, λέει και αυτά τα μέτρα της Τουρκίας τα οποία δεν συνάδουν προς αυτή την Τελωνική Ένωση. Άρα θα πρέπει η Τουρκία να κάνει τα βήματα που χρειάζονται τόσο ώστε να λειτουργήσει η Τελωνική Ένωση και να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικές συμφωνίες τους ώστε οι οικονομικές μας σχέσεις να αναβαθμιστούν επίσης με την ευκαιρία θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεσμεύομαι να βοηθήσω τη σύσφυξη των σχέσεων με την Τουρκία. Τηλεφώνησε ο Τούρκος υπουργό Εμπορίου και κανονίσαμε να συναντηθούμε Του άμεσους μήνες με προσεκάλεσε, αποδέχεται την πρόσκληση, ούτως ώστε να δούμε πώς θα προοδεύσουν οι σχέσεις μας και πώς με φιλικό τρόπο και επικοδομητικό θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα σε εμπορικέ μα σχέσει. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, και τώρα οι των πολιτικών ομάδων και ξεκινούμε με την κυρία Τρόβολ. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βεβαίως έναν ε, ισχυρό οικονομικό εταίρο στο πρόσωπο της Τουρκίας ε, και αντιστρόφως παρά το ότι βεβαίως έχει διαφοροποιηθεί έχουν διαφοροποιηθεί τελευταία οι εμπορικές ροές της εξακολουθούμε να είμαστε ο μεγαλύτερος εταίρος της ε, Τουρκίας βεβαίως ε, μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα όπως αναφέρει και η έκθεση παραδείγματος χάρη ζητάμε να μειωθούν οι υψηλοί δασμοί στα αγροτικά προϊόντα και να σταματήσουν οι, τα μη δασμολογικά εμπόδια και κυρίως να υπάρξει μία απλοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας η οποία θα βελτιώνει το εμπόριο. Βεβαίως υπάρχουν και βελτιώσεις ε, που επέφερε τελευταία η Τουρκία, τις ανέφερε ο κύριος Επίτροπος παρόλα αυτά οι ξένες επενδύσεις θα ήταν μεγαλύτερες εάν ήταν δυνατόν να βελτιωθεί η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και να τήρει τους κανόνες η Τουρκία καθώς δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι νόμοι στην Τουρκία. Πρέπει επίσης να ζητήσουμε από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Τήθες Σύνδεσης. Εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών που πρέπει να σταματήσουν. Μια τελευταία πρόταση. Όταν μιλάμε για την ε, Τουρκία και στην Επιτροπή Εμπορίου πάρα πολύ συχνά μιλάμε με έντονα συναισθήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, εισηγητή γιατί κατάφερε σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο μας εκφράζει όλους, κάτι το οποίο έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Καζακ, ευχαριστώ κύριε Ρόβολ, η κυρία Μπαλτσάνη για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν εμποδι... βαθιές εμπορικές σχέσεις. Η Τελωνιακή Ένωση επέτρεψε να, φτάσει, να φτάσουν οι εμπορικέ ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών το 100 δις το χρόνο. Ιδίως ωστόσο η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας την καθιστά εξαιρετικά σημαντικό ε, σημείο σύνδεσης της ε, περιοχής Μεσογείου, ε, Ευξήνου Πόντου, Καυκάσου, Μέση Ανατολής. Η Τουρκία ε, είναι αντίθετη, έχει αντίθετη πορεία από την Ευρώπη. Είναι μια δυναμική κοινωνία με νέο πληθυσμό που πρώτη αντιμετώπισε την κρίση και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Είναι λοιπόν μια χώρα συμπληρωματική διότι διαφορετική από πολλές οπτικές γωνίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την οποία οποία υπάρχουν κατά συνέπεια μεγάλες δυνατότητες ένθεν κακήθεν. Και από αυτού πρέπει να, να στραφούμε ιδίω, να προσέξουμε, να μην διασπαθήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, να προωθήσουμε καρποφόρες επενδύσεις. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικός εμπορικός εταίρος. Η Τουρκία, ωστόσο, προσβλέπει όλο ένα και περισσότερο προς τη Ρωσία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή. Η Τελωνιακή Ένωση δεν εφαρμόζεται ακόμα στις δημόσιες αγορές, δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες. Παραμένουν λοιπόν μεγάλα εμπόδια ακόμα για το διεθνές εμπόδιο. Κατά συνέπεια πρέπει να δουλέψουμε για να αφαιρέσουμε τους φραγμούς και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και προς τα εκεί πηγαίνει η έκθεση που συζητούμε και θα ψηφίσουμε τις επόμενες ημέρες. Διότι υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται πραγματικά να αυξηθούν οι δυνατότητες, η, ενέργεια, το περιβάλλον, οι υπηρεσίες, οι υποδομές. Και για τις σχέσεις αυτές, για να μπορέσουν οι σχέσεις αυτές να προχωρήσουν, πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την έκθεση του κυρίου Καζάκ που τον ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχει καταβάλει. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλτη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε, αγαπητέ κύριε επίτροπε, χαίρο είμαι ευχαριστημένος από την έκθεση Καζάκ που μας λέει κατά βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω στις πολιτικές και άλλες σχέσεις με την Τουρκία. Ιδίω στην εμπορική πολιτική. Υπενθυμίσαμε ήδη την κρίσιμη στρατηγική θέση τη Τουρκία εναντί τη Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή, τη Κεντρική Ασία και του Καυκάσιου. Υπάρχει ένα ποίημα του Χικμέτ, του Αζίν Χικμέτ, που λέει ότι αυτή η χώρα που μοιάζει με ένα κεφάλι από μία, ε, από μία φοράδα που έφτασε και έκατσε και για να πιει νερό στη Μεσόγειο. Αυτή το δείχνει το κομβικό σημείο της Τουρκίας για το, την περιοχή αυτή που είναι ένα κέντρο. Για το σκοπό αυτό ωστόσο θα πρέπει να στεφεροποιηθούν οι πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με την Αρμενία, να κλείσει το Κυπριακό και θυμίζω την παράγραφο 11 της έκθεσης Καζάκ για την εφαρμογή της Τελωνιακής Ένωσης και το τμήμα της Κύπρου που κατέχει, που είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας, δεν τα θύμισε όλα η κυρία Μπαλτζάνη. Υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα στην, παρα, στην παραποίηση, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην ε, εφαρμογή της Τελωνιακής Ένωσης των τομέα των υπηρεσιών και των ε, διαγωνισμών. Ευχαριστώ ωστόσο τον κύριο Καζάκ. Η Μεσόγειο θα αλλάξει και, θέλει, και θέλουμε να αλλάξουμε μαζί με την Τουρκία η ανάπτυξη της οποίας για το 2000, μέχρι το 2020 προβλέπεται να φτάσει το ποσοστό του 37%. Αυτό μας λέει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φινάλντι. Η κυρία Κέλλαρη για τους πράσινους ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή για την καλή σας έκθεση, η οποία νομίζω δείχνει πόσο σημαντικός εμπορικός εταίρος είναι η Τουρκία για την Ένωση και αντιστρόφως και πόσο σημαντική είναι η Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα και στις δύο πλευρές και στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Τουρκία παραδείγματο χάρη πρέπει να ενισχυθούν μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που πρέπει να δούμε στην Ένωση, ένα από τα οποία είναι απελευθέρωση της βίζας. Δεν πρέπει να απελευθερώνουμε μόνο την θεώρηση για οδηγούς φορτηγών και επιχειρηματίες, αλλά και για φοιτητές, τουρίστες, για να ενισχυθούν οι σχέσεις και μεταξύ των κρατών και μεταξύ των ανθρώπων. Όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρω εμπορίου, πρέπει να εμπλακεί πλήρω η Τουρκία στη διαπραγματεύση, εφόσον βεβαίως επηρεάζεται και ολοκληρωτικά. Σε γενικές γραμμές η σχέση μας πρέπει να είναι δίκαιη και αυτό συμπεριλαμβάνει την ξεκάθαρη δήλωση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τις υποσχέσεις της και θα καλωσορίσει την Τουρκία ως μέλος μόλις εκπληρωθούν τα κριτήρια της Κομεχάγης. Σας ευχαριστώ για την ΓΚΟΕ ο κύριος Τριανταφυλλίδης για 1,5 λεπτό. Το δημοψήφισμα για τις συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία είχε θετική έκβαση αλλά αποτελεί μονάχα ένα μικρό βήμα προ την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατομικών πολιτικών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Μέρο των κούρδων και άλλων απήχαν από την ψηφοφορία ή καταψήφισαν ακριβώς επειδή απαιτούνται βαθύτερες βελτιώσεις και αυτονόητα δικαιώματα. είναι λυπηρό το ότι δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί νομοθεσία κατά τα πρότυπα της διεθνούς οργάνωσης εργασίας η καταψηφισαν ακριβω επειδη απαιτουνται βαθυτερε βελτιωσει εισάγει τον πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα τη διεθνου οργανωση εργασια η οποια να οργάνωσης τη απεργία και τη συλλογική διαπραγματεύση ω πολιτική ομάδα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η πρόοδο δεν μετριέται μόνο από το εμπόριο και τι οικονομικέ σχέσει μια χώρα. χαιρετίζουμε το γεγονό ότι και μέσα από αυτή την έκθεση το ευρωκοινοβούλιο στέλνει στην τουρκία ένα σταθερό μήνυμα δεν είναι αποδεκτή η επιλεκτική εφαρμογή ή καλύτερα η μη εφαρμογή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας χωρίς να υπάρξουν σοβαρέ επιπτώσει στι ενταξιακέ διαπραγματεύσεις γι' αυτό εάν η τουρκία επιθυμεί το εμπόριο της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την ευρωπαϊκή ένωση αντί να ψάχνει για έμμεσους τρόπους αναγνώρισης μιας οντότητας που βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του οργανισμού ηνωμένων εθνών είναι παράνομη ας αποδεχτεί την πρόταση του προέδρου της κυπριακής δημοκρατίας δημήτρη χριστόφια να επιστρέψει μέσω του οηε την αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της και να τεθεί το εμπόριο στο λιμάνι της πόλης αυτής υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής ένωσης. αφού αυτή η πρόταση μη ενέχοντα καμιά σκοπιμότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση τη τουρκοκυπριακής κοινότητα και ταυτόχρονα να αποτελέσει πεδίο εμβάθυνση των προσπαθειών επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων στο νησί. Ευχαριστώ. για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της δημοκρατία ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση περιγράφει την Τουρκία ως την έκτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Ε, αντικειμενικά μιλώντας, ε, η έκταση της χώρας που λέγεται Τουρκία είναι πάνω από 300.000 τετραγωνικά μίλια. Από αυτά, μόλις 3,5% βρίσκεται στην Ευρώπη. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κατατάξει την Τουρκία στην Ευρώπη. Από το 1995 έχουμε τελωνιακή ένωση με την Τουρκία. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Το Μονακό και η Ανδόρα είναι οι μόνες άλλες χώρες ε, που έχουν κάτι τέτοιο. Να έρθω σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Η ύπαρξη και η επιτυχία της Τελωνιακής Ένωσης κάνει το να καταστεί η Τουρκία πλήρες μέλος με ό,τι σημαίνει αυτό κάτι το τελείως περιττό Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητάμε στην Ευρώπη για αρκετό καιρό ακόμα. Σας ευχαριστώ η κυρία Στάσεν για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μπροστά μας την έκθεση για το ελεύθερο εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Από το 1996 που έχουμε τελωνιακή ένωση με την Τουρκία έχουμε ισχυρό και υψηλό εμπόριο. Και βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε θετικό και θα πρέπει πράγματι να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια και τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Το ελεύθερο εμπόριο είναι καλό για όλους μας και για τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Τουρκία. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι ξεκάθαρο πω εμείς θεωρούμε πως εκεί πρέπει να σταματήσουν οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Είμαστε ως κόμμα για την ελευθερία κατά της ε, ένταξης της Τουρκίας. Μπορεί να είναι μια μεγάλη χώρα με την οποία έχουμε βεβαίω ε, εμπορικέ σχέσει. Εμπορικέ σχέσει έχουμε με τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία, πολλέ άλλε χώρε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και αυτέ ε, κράτη-μέλη. Ω εμπορικό εταίρο, πράγματι αυτό δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό ω κόμμα. Αλλά το να γίνει η Τουρκία μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Αυτό κατηγορηματικά όχι. Σα ευχαριστώ, η κυρία Ομουν κατόπιν. Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια Τουρκίας για το Κοινοβούλιο θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή αυτή της έκθεσης. Σύμφωνο μαζί του πως η Τελωνιακή Ένωση έχει πολλά θετικά αποτελέσματα και για Τούρκους και για Ευρωπαίους επιχειρηματίες αλλά όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος η Τελωνιακή Ένωση σε πολλά σημεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ευκαιρίε και οι προκλήσεις για τις εμπορικές μας σχέσεις με την Τουρκία είναι σαφείς. Τα εμπορικά εμπόδια και τα τεχνικά εμπόδια τα οποία εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν πρέπει γρήγορα να παραμεριστούν και βεβαίως θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε περαιτέρω εναρμόνιση όταν προχωρήσουμε παραπεραστό και εκτιμένο. αλλά θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει κάποια καταπολέμηση της πειρατείας των προϊόντων. Γιατί πάρα πολλέ ευρωπαϊκές μάρκες και πάρα πολλοί ευρωπαίοι κατασκευαστές υποφέρουν από απομιμήσεις προϊόντων, ε, παιχνιδιών, ε, που τα παιχνίδια ε, σημαίνουν και κινδύνους και για τους Τούρκους πολίτες. Επίσης θεωρώ σημαντικό να σταθούμε στο σημείο της κοινωνικής οικονομίας και συγκεκριμένα τώρα που εγκρίθηκε το που πέρασε το δημοψήφισμα να συζητήσουμε και για τα συνδικάτα και για το πώς θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Κύριε Πρόεδρε, επίσης στην ενέργεια έχουμε κοινά συμφέροντα. Πρέπει, πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε εδώ πέρα. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, συχνά διαπιστώνω πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα γιατί ε, υφίστανται διαφορετική μεταχείριση και θα τα πω αυτά στον κύριο Επίτροπο. Όμως κρίσιμο για την Τουρκία παραμένει βεβαίως ε, η πλήρης εφαρμογή του ε, προσθέτου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εάν συμβεί αυτό, εάν κυρωθεί αυτό κύριε Πρόεδρε, τότε θα έχει φύγει από τη μέση ένα τεράστιο εμπόδιο για τις περαιτέρω σχέσεις και εμπορικές ε, σχέσεις ε, και βεβαίως ε, από αυτό θα επωφεληθεί και η Τουρκία και η Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως καλό είναι το ότι έχουμε αυτή την έκθεση τώρα και βεβαίως τα πολιτικά ζητήματα θα τα δούμε στην επόμενη έκθεση την οποία θα συζητήσει η Επιτροπή Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αρίφ είναι επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα, θα ήθελα να σας πω μια γενική παρατήρηση για την έκθεση. Γιατί ε, τις σχέση μας με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει ε, οι ειδικέ και σκιώδες και να του συγχωρείτε. Δηλαδή, θέλω να πω, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ε, θολή αυτή η έκθεση σε σχέση με, και, και διαφορούμε οι σχέσει μα, γιατί έχουμε τι θέσει τη Κοινοβουλική Επιτροπή και το θέμα το, το οποίο διαπνεί όλε αυτέ τι σχέσει και είναι κάτι που βρίσκεται πέρα από τι οικονομικέ σχέσει με την Τουρκία. Και είναι αυτό κάτι που αναφύγεται συνέχεια υπέρ ή κατά τη προσχώρηση είμαστε προσφόρηση της Τουρκίας Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το κρίνουμε σε σχέση με, την Τουρκία. Σαν ήταν μια οποιαδήποτε χώρα, γιατί θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικέ σχέσει, είναι υποψήφια χώρα και γι' αυτό το λόγο έχει κάποιε συγκεκριμένε υποχρεώσει που θα πρέπει να εκτελέσει και αυτή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι δύσκολο να πούμε κατά πόσον αυτή η έκθεση δικοτουρίζει τι σχέσει με την χώρα και κατά πόσον έτσι μπορεί να μας βοηθήσει να χαράξουμε τη στρατηγική. Θα πρέπει να δούμε ε, αν είμαστε για το ναι ή για το όχι. Θέλουμε να είναι προμήγο εταίρος ή θέλουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να πούμε προσοχή, προσοχή για αυτή την αντίφαση ότι δεν μπορεί από μια μεριά να είμαστε τόσο διαφορούμενοι για τον κοινό προορισμό και από την άλλη μεριά να θέλουμε να έχουμε την Τουρκία σε κάποιες αποστάσεις γιατί εταιρικέ σχέσεις σημαίνουν ειλικρίνεια, σημαίνουν εμπιστοσύνη γιατί βέβαια θα πρέπει η Τουρκία να καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε, ούτω ώστε να τι υποχρεώσει, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει από τη μεριά μα να δείξουμε ενθάρρυνση, να δείξουμε εμπιστοσύνη ε, και να στείλουμε κάποια θετικά μηνύματα. Και προσπαθούν να κάνουν αυτά που ζητούμε, σιγά σιγά συντονίζουν το δίκαιό του με τα δικά μας κριτήρια για να γίνουν πλήρες μέλος, ακόμα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, πολλές προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να μην τους βάζουμε πλέον ε, φραγμούς και να μην εμποδίζουμε τις σχέσεις αυτές να οδηγήσουν στην προσχώρηση. Βλέπω μία μπλε κάρτα, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Έχω μια ερώτηση να υποβάλω. Ο αγορητής ξέρει ότι αυτό το σύνταγμα το οποίο ψηφίστηκε υπονομεύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και συμφωνείτε με αυτό. Ξαφίσταν η ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε. Βεβαίω έχουμε τα πέρα και τα κατά, είναι περίπλοκη αυτή η μεταρρύθμιση. Τώρα είναι λιγότερο, προχωρεί η δημοκρατία, είναι λιγότερο σημαντικό ο στρατό. Προχωρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε μπορούμε να βρούμε τέτοιε κατηγορίε ε, για τα πράγματα που δεν είναι τέλεια. Εγώ όμω ε, από τη φύση μου δεν είμαι απεσιόδοξο. Επομένω νομίζω ότι ό,τι κινήσει κάνει η Τουρκία μα σωστή κατεύθυνση και ότι θέλουν να, ε, να, να προσχωρήσουν, επομένω και εμεί να του βοηθήσουμε. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Κυρία, Κύριε Γέτεν Μάκη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κύριο Καζάκ. Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή και αντίθετα από τον κύριο Αρίφ, τον προηγούμενο μιλητή, εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να καλύψουμε τα πάντα εδώ. Η έκθεση είναι μια έκθεση για, εμπορικούς, ε, για εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Ένα από το, τα προβλήματα του Κοινοβουλίου είναι ότι κάθε φορά που εμφανίζεται μια έκθεση βάζουμε τα πάντα σε αυτήν και τελικά δεν λέμε τίποτα το ουσιαστικό. Η έκθεση ασχολείται με τα βασικά ζητήματα και ευχαριστώ τον εισηγητή γι' αυτόν. Το 1996 η Τελωνική Ένωση μεταξύ Ευρώπης και Τουρκία έφερε την Τουρκία πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός εταίρος με όλες τις χώρες της Ένωσης και με την Ένωση. Δυστυχώς, ωστόσο, η Τελωνιακή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, ε, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων. Οι τουρκικές αρχές ζητούν άδεια, ζητούν άδεια να υπάρχουν άδειε σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αντιβαίνει στην Τελωνιακή Ένωση. Και οι ευρωπαϊκέ χώρε το κάνουν, αλλά πρέπει να αναλάβουμε από κοινού δράση. Ο εισηγητή μίλησε για τα προβλήματα των προϊόντων απομίμηση. Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά στον τομέα αυτό. Και βεβαίω ένα από τα σοβαρά προβλήματα στην Τουρκία είναι η αφανής οικονομία που καλύπτει ένα τερά, μεγάλο ποσοστό της οικονομίας ε, και έχει μεγάλες επιπτώσεις στο εμπόριο και στην οικονομία της χώρας. Οι μελλοντικέ εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα αυτό, να λειτουργήσει σωστότερα η Τελωνιακή Ένωση σε κάθε επίπεδο. Η κυρία Τζαφέλ, επόμενη ομιλήτρια, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να προσθέσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην αντικειμενική έκθεση του κυρίου καζακ και επιτρέψτε με να κάνω δύο παρατηρήσεις με ρεαλισμό. η πρώτη αφορά την παράγραφο 26 για τον ενεργειακό εφοδιασμό. πιστεύω ότι και η επιτροπή και το ευρωκοινοβούλιο έχει υπερεκτιμήσει την σημασία της τουρκίας για τον ενεργειακό τομέα. η τουρκία δεν παράγει ενέργεια. η τουρκία είναι μια εξαιρετική δίοδος για ενεργειακά δίκτυα. δεν μας λύνει ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν και άλλα δίκτυα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η μεταφορά της ενέργειας. ας είμαστε ρεαλιστές και ας δούμε ότι στον ενεργειακό τομέα όλα αυτά που συζητάμε ναμπούκο και τα λοιπά και όλα αυτά είναι ασκήσεις επιχάρτου γιατί η ίδια η χώρα η τουρκία δεν μπορεί να μας προμηθεύσει ενέργεια. αντιθέτως είναι μια χώρα με μεγάλη βιομηχανία η οποία χρειάζεται ενέργεια και θα πρέπει να τη βλέπουμε έτσι. δεύτερο σημείο που θέλω να τοποθετηθώ επειδή μιλάμε για εμπόριο δεν μπορεί να αναφερόμαστε στο άνοιγμα εμπορίου με την τουρκία όταν στην τουρκία ανθεί η αγορά της παραγωγής ε, απομιμήσεων ευρωπαϊκών προϊόντων. κύριε πρόεδρε όπου και να πάτε σε βιτρίνες ανοιχτά σε τουρκικά παζάρια είναι γεμάτα με πολύ καλές ομολογουμένως απομιμήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων. Αν είναι δε και είσοδος απομιμήσεων από την ανατολή. αν δεν λύσουμε τα προβλήματα εμπορίου που έχουμε με την τουρκία που πλήττουν την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έχετε χρόνο. να συζητάμε άλλα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Παπαστάμκος, επόμενος ομιλητής. 1,5 λεπτό. Ε, αναγνωρίζουμε τη σημασία των εμπορικών σχέσεων Ένωσης Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τήρησε υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην εξισορρόπηση του αρχικού κειμένου της συζητούμενης έκθεσης. Καλούμε την Τουρκία να εκπληρώσει πλήρως και αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις και υπενθυμίζουμε ότι η σχετική παράληψη ενδέχεται να επηρεάσει ακόμα πιο σοβαρά την πορεία των διαπραγματεύσεων θα ήθελα και εγώ να επισημάνω αυτό που και ο κύριος ρινάλντι αλλά και μόλις ε, τώρα η κυρία τζαβέλα ε, τόνισαν ότι η τουρκία διατηρεί υψηλή θέση μεταξύ των χωρών που παράγουν προϊόντα απομίμησης και κατάσχονται στην εε επαναλαμβάνω υψηλότατη θέση και ότι δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. η εξωτερική δράση της ένωσης κυρίες και κύριοι συνάδελφοι περιλαμβανομένης της ε, κοινή εμπορικής πολιτικής επιδιώκει τη διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής και το σεβασμό των αρχών του καταστατικού χάρτη των ηνωμένων εθνών και του διεθνούς δικαίου καθώς και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις ανωτέρω αρχές. εκπτώσεις αυτής της θεμελιώδους διακηρυκτικής αρχής της συνθήκης της λισαβόνας δεν νοούνται. και να έχουμε πάντα προοφθαλμόν ότι δεν διαπραγματεύεται η ευρωπαϊκή ένωση με την τουρκία αλλά η τουρκία με την ευρωπαϊκή ένωση για την προσχώρησή της και το βάρος της προσαρμογής βαρύνει την ίδια την τουρκία. όπερ έδι δείξε. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Thank you. Our next speaker is Mr. Ο κύριος Κούτας, επόμενος μιλής, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Τουρκία είναι η έβδομη εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μόνη χώρα υποψήφια για ένωση που έχει τελωνική ένωση με την ΕΕ. Πρόκειται λοιπόν για μια προνομιούχα σχέση όπου η ανταλλαγή, οι εμπορικές και οικονομικές αναλλαγές παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταίροι πρέπει να συνεργαστούν για να ευθυγραμμίσουν τις εμπορικές πολιτικές τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με τρίτε χώρες. Η Τελωνική Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί με την υλοποίηση ασφαλών προβλέψεων για τις δημόσιες αγορές και τις υπηρεσίες, ενώ πρέπει να βρεθεί και μία λύση για το ζήτημα των θεωρήσεων, ούτω ώστε να μπορούν οι Τούρκοι επιχειρηματίες να εισέλθουν στην Ένωση. Χρειάζεται η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών να γίνουν πιο στενές και να δώσουμε σαν Ένωση μια ε, σαφέστερη προοπτική στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που διαπραγματεύεται εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι οι διαπραγματεύσεις ε, μακροσκελέστατες ε, καθώς για λόγους πολιτισμού και παράδοσης απέχει πολύ από την Ευρώπη η Τουρκία. Βεβαίως οι επιχειρηματικές σχέσεις μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία, την συνεργασία στο μη εκείνους όπου οι Τούρκοι πολίτες βρίσκουν κάποιο κοινό έδαφος με τους Ευρωπαίους και υπάρχει βεβαίως και αμοιβαίο συμφέρον. Με βάση αυτά μετά μπορούμε να οικοδομήσουμε μια φιλία και αμοιβαία εμπιστοσύνη και να μιλήσουμε ανοιχτά με τους Τούρκους φίλους μας για τα προβλήματα που μας ανησυχούν γιατί είμαστε γείτονες και εταίροι της Τουρκίας. Πρέπει να εξηγήσουμε ξεκάθαρα πως ε, οποιοδήποτε φέρνει παραποιημένα προϊόντα στην αγορά δεν είναι παρακλέφτης γιατί κλέβει ξεκάθαρα από ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει επίσης να εξηγήσουμε πως η Τελωνιακή Ένωση δεν ε, είναι χώρος για να κάνει κανείς τον έξυπνο και να βάζει τεχνικά ε, δασμολογικά εμπόδια. Πρέπει να διδάξουμε στους Τούρκους φίλους μας να συμπεριφέρονται πολιτισμένα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριος Βαλέσα να ευχαριστήσω τον κύριο Καζάκ, τον συντάκτη τη έκθεσης γιατί προσπάθησε να γράψει μια μερόληπτη έκθεση για τι εμπορικέ σχέσει με την Τουρκία. Τα πιο επίμαχα σημεία, η αρνητική πλευρά των χρησιών μας, καλύπτω την έκθεση, επομένω η έκθεση είναι αξιόλογη. Το πιο σημαντικό είναι θα πρέπει να συνεχίσει η Τουρκία τις προσαρμογές ως αυτό το εμπορικό δίκαιο για να συνάδει προς τις Ευρωπαϊκές Ένωση, επομένω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτές τις, ε, τα κίνητρα που υπάρχουν ή τα αντικίνητρα για ξένους επενδυτές, επενδυτές ε, γραφειοκρατία, δασμοί, δύσκολη, συνεργασία. Άρα μόνο εάν έχουμε πλήρη εφαρμογή των όσων πρέπει θα έχουμε καλή συνεργασία και θα ευοδοθεί η διαδικασία της ένταξης. Ελπίζουμε αυτή η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επιτυχής. Η κυρία Μπιζότο, ένα λεπτό. Είναι προφανέ θετικό να εμβαθύνουμε σαν Ευρώπη τι σχέσει μα με γειτονικέ χώρε. Ωστόσο, η Ένωση μέχρι τώρα είχε μια εμπορική πολιτική κατά τον τρίτο χρόνο, πάντα υπόψη και κοινωνικέ και ανθρωπιστικέ διαστάσει. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμιστεί η διάσταση αυτή με αποφασιστικό τρόπο και έναντι της Τουρκίας, μιας χώρας η οποία γίνεται όλο και πιο ισλαμική και όπου η θέση της γυναίκας επιδεινώνεται με πάνω από 1500 γυναίκες που θανατώθηκαν το 2009 σε ε, βία στο σπίτι. Μια χώρα όπου οι χριστιανοί ζουν υπό τον κίνδυνο των επιθέσεων από Ισλαμιστές. Ε, η, η δολοφονία του, του Βανέζε ε, το δείχνει. Η Τουρκία πρέπει να προωθήσει ταυτόχρονα και να δείξει ότι προωθεί μια δίκη, ένα δίκαιο εμπόριο. Ένα πράγμα που είναι βέβαιο είναι ότι πρέπει να ε, ανησυχήσουμε για τον ε, ρόλο πολιτική καθοδήγηση που προσπαθεί η Τουρκία να αποκτήσει στον Αραβικό κόμμα, τι σχέσει κόσμο, τι σχέσει που έχει με το Ιράν και την υποστήριξή τη Ναμά. Η εμπορική πολιτική πρέπει να υπάρχει βεβαίω, αλλά αυτή δεν πρέπει να γίνει δούριο ύπο για να διευκολυνθεί η ένταξη τη Τουρκία στην Ευρώπη. Κέστιγκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν πολύ καλές οικονομικές σχέσεις και οπωσδήποτε πρέπει να επεκταθεί το εμπόριο με την Τουρκία για να έχουμε αφενός οικονομική ανάπτυξη και στις δύο πλευρές και στην Ένωση και στην Τουρκία για έτσι. Καλώς ορίζω την έκθεση πρωτοβουλίας αυτή η οποία βέβαια τονίζει αρκετά ζητήματα, έστω και αν δεν είναι πάντα θετικά αυτά. Βλέπουμε Παραδείγματο χάρη την πειρατεία προϊόντων, ε, εμπόδια που υπάρχουν σε φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και σε ζητήματα δημοσίων προμηθειών. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, διατάξεις εκείνες οι οποίες ε, είναι προστατευτικές όσον αφορά το εμπόριο για τα γεωργικά προϊόντα μιλάμε για ένα ποσοστό απασχόληση στον γεωργικό τομέα άνω του 26% στην ε, Τουρκία, οπότε λογικό είναι να αποδίδουν σε αυτό μεγάλη σημασία. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνει εις βάρος των ευρωπαϊκών γεωργικών επιχειρήσεων και εις βάρος και σε αντίθεση με την νομοθεσία της Ελληνιακής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να καταργηθούν το συντομότερο δυνατό αυτά τα εμπόδια. Δεν είναι δυνατόν τα υψηλά ποιοτικά προϊόντα της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν άδικα εμπόδια. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στη δικασία του KTI. Βλέπω την κυρία Γιάς Λοβιέτσκα, οπότε θα της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια με καλές στιγμές και κακές. Πάρα πολύ καλά τα αποτυπώνει ο κ. Χαζάκη στην ε, έκθεση, όμω ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή τη Τελωνική Ένωση για διάφορου λόγου που οφείλονται στου μεν και στου δε. Και πάντω η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παράγων στην ευρύτερη περιοχή. Ε, αλλιώς, ε, αν δεν πλησιάσουμε την Τουρκία, δεν θα φέρουμε σταθεροποίηση στην Μέση Ανατολή, δεν θα έχουμε κάποια επιρροή στα της ε, ε, αγοράς και φυσικού αερίου. Άρα να λάβουμε υπόψη μα και το ρόλο στη Μέση Ανατολή τη χώρα εκείνα και αν δεν το προσέξουμε αυτό, δεν προσέξουμε τι εμπορικέ σχέσει, τότε στο τέλο θα βγούμε, θα μην θα χάσουμε την Τουρκία όπω χάσαμε την Αφρική. Η τουρκική κοινωνία κρύωσε. Ε, και, και το λέω διπλωματικά, τουλάχιστον έχει κρυώσει όσον αφορά τη ζέση της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς να βαθμίσουμε σχέση με τη χώρα αυτή. Now Mr. has the floor. Ο κύριο Πάσκου. Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία είναι, έχουν και πολιτική διάσταση. Παρότι αναγνωρίζει το γεγονός αυτό ωστόσο, η Ένωση δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποφύγει την εντύπωση ότι ε, παίζει ένα παιχνίδι όποιο κλείσει πρώτο τα βλέφαρά του με την Τουρκία η Τουρκία περιμένει να διακόψει η Ευρώπη περιμένει η Τουρκία να διακόψει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξαντλημένη από τις ε, ε, Αναβολέ. Δυστυχώ ε, το καλά νέα είναι ότι με τα τελευταία δεδομένα η Τουρκία είναι ε, απογοητευμένοι από την Ένωση και παρότι η Ένωση είναι ο κύριος εταίρος της Τουρκίας αρχίζει και την προλαβαίνουν, την προλαβαίνουν άλλες χώρες, αραβικές χώρες, Ρωσία κλπ. Δεν πρέπει η έκθεση αυτή να μας κάνει να αγνοήσουμε το βασικό μας ζήτημα είναι να αποφασίσουμε ή όχι κατά πόσον θέλουμε ή όχι την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση. Ε, σίγου, σίγουρα δεν μπορούμε να Είμαστε αντίθετοι με μια περαιτέρω φιλελευθερωποίηση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το κόστο εργασία στην ε, Τουρκία είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι για μα. Αν ανοίξουμε λοιπόν τα σύνορα μα, σημαίνει ότι, επιβλα... ότι βλάπτουμε την ευρωπαϊκή αγορά και ε, ενισχύουμε την... τον αθέμητο ανταγωνισμό. Η απλοποίηση των εμπορικών ανταλλαγών με την Τουρκία είναι λάθο, κατά την άποψή μου. Ε, πιστεύουμε ότι το σύστημα, το κοινωνικό, πολιτικό και ε, ε, κοινωνικό σύστημα είναι μακρά από εμά. Και η θρησκεία ακόμα είναι διαφορετική. Το να είσαι χριστιανός στην Τουρκία σημαίνει ότι βρίσκεσαι, ότι αντιμετωπίζει κίνδυνος. Το να ο Ισλαμισμός γίνεται ο κανόνας παντού στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις μας δορίζοντας στην Τουρκία απλοποίηση εμπορικών ανταλλαγών με τη χώρα μας. Με τις χώρες μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητάμε εδώ μέσα για λειτουργικές εμπορικές σχέσεις και για βελτίωση της Ελληνιακής Ένωσης με την Τουρκία, αυτό βεβαίως είναι κομμάτι της διαδικασίας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον προς τα εκεί θα έπρεπε να οδηγήσει. Επίσης γνωρίζουμε πως οι κριτικοί αυτής της ένταξης μιλάνε πάντα για μια προνομιακή σχέση ως εναλλακτική και Ε, βεβαίως ε, λόγος είναι πως ε, ήδη υπάρχει μια τέτοια προνομιακή σχέση. Θα πρέπει όμως να την δικαιολογήσει και να την κερδίσει και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στο πολιτικό επίπεδο. Αν δούμε το τι γίνεται με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, το ότι ε, αρνείται να επιλύσει σε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση το Κυπριακό, όπως υπάρχει ακόμα διακριτική μεταχείριση των Κούρδων, αντιλαμβάνεται πως Μόνο με τι εμπορικέ σχέσεις δεν υπάρχει ξευρωπαϊσμό τη Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. 12 Acesta demonstrează turce față de regimul democratic, singurul acceptabil în Europa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 Πρόεδρε, η Τουρκία έχει υποφεληθεί από την πολύχρονη τελωνιακή τη σχέση. Ωστόσο, η τελωνιακή σχέση για να καταστεί ακόμη πιο λειτουργική χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση πολλών εκκρεμούν των θεμάτων. Η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίσει καλύτερα τι εμπορικέ τη πολιτικέ και το περιφερειακό εμπόριο, να μειώσει τη γραφειοκρατία, τα προϊόντα απομίμηση, τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδικαλιστών και μειονοτήτων, να αντιμετωπίσει το χαμηλό επίπεδο συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασία, να προωθήσει τη την νεανική απασχόληση. κυρίω οφείλει να εφαρμόσει πλήρω το πρόσθετο πρωτόκολλο τη συμφωνία σύνδεση να άρει το εμπάρκο σε βάρο κυπριακών πλοίων και αεροσκαφών να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο και να σεβαστεί τι συμβάσει τη διεθνού οργάνωση εργασία όσον αφορά το συνδικαλισμό το δικαίωμα στην απεργία και στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. ευχαριστώ. Τελευταίος, αλλά σημαντικός, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον ε, κύριο Καζάκ για μια πολύ καλή και αντικειμενική έκθεση. Πράγματι, οι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντικέ και γι' αυτό πρέπει να τι προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά πρέπει και να αναδεικνύουμε τα σημεία στα οποία επιδέχονται βελτίωση πρέπει να σας πω λοιπόν να αναφερθώ σε δύο από αυτά τα σημεία. θεωρούσαμε και υπάρχει συζήτηση κατά πόσον η τουρκία είναι μια ευρωπαϊκή ή μη ευρωπαϊκή χώρα. εμείς σίγουρα θέλουμε την τουρκία μια ευρωπαϊκή χώρα και να μπορέσει να γίνει κάποτε μέλος της οικογένειας. όμως όσον αφορά τα πειρατικά προϊόντα τα προϊόντα απομίμησης και την μη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων η τουρκία είναι σίγουρα περισσότερο ασιατική παρά ευρωπαϊκή χώρα το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά την τελωνειακή ένωση κύριε πρόεδρε. η τελωνειακή ένωση είναι ο πυρήνας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. δεν είναι λοιπόν νοητό μια υποψήφια χώρα να μην έχει εφαρμόσει στην πλήρη εφαρμογή του την τελωνειακή ένωση και να υπάρχει κράτος μέλος με το οποίο η τουρκία αρνείται να προχωρήσει σε τελωνειακή ένωση και αυτό το κράτος μέλος είναι η κυπριακή δημοκρατία. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Επιτροπής ο κύριος ε, Ντεούτ για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είναι σαφές από τις παρεμβάσεις πως υπάρχει συνένεση όσον αφορά την έκθεση και θα ήθελα να πω λίγα λόγια για κάποια ζητήματα, για τα, ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία με συμφωνία συμφωνίες ελευθερού εμπορίου με του εταίρους στην Ευρώπη, το ζήτημα της βίζας και την επιβολή νομοθεσίας ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί πράγματι η πνευματική ιδιοκτησία και η πειρατεία αναφέρθηκαν κάτω επανάληψη. Επίσης, ανησυχώ, και η Κομισιόν θα συνεχίσει να πιέζει για αυτά τα ζητήματα. Μετά από χρόνια επανειλημμένων ετοιμάτων δέχτηκε η Τουρκία πρόσφατα να συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Πρόκειται για ένα πρωτοθετικό βήμα και ελπίζω η ομάδα αυτή εργασίας να μας βοηθήσει να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Δεύτερον, για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στην σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Η Τουρκία εδώ και χρόνια λέει πως υφίσταται επιπτώσεις λόγω της ε, δυσκολίας ε, του να συνάψει συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με κάποιους εταίρους της Ένωσης. Βεβαίως ο αριθμός των κρισίμων αυτών συμφωνιών είναι περιορισμένος. Επίσης η Τουρκία δεν έχει υποβάλει παρά τα αιτήματα της Κομισιόν δεδομένα για τα συνέπειες αυτές οι οποίες επικαλείται. Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε πως η Κομισιόν δρά πλήρως εντός των συμφωνιών Τελωνιακής Ένωσης και μάλιστα προχώρησε και πέρα από τις υποχρεώσεις της ε, βοηθώντας ε, την ε, Τουρκία με το να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τους εταίρους μας με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει ελευθερία και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίω, ε, το να προσκαλέσουμε την Τουρκία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με του εταίρου αυτού, αυτό είναι κάτι το τελείω διαφορετικό. Τώρα, για τα ζητήματα βίζα αυτά δεν καλύπτονται από την Ελληνική Ένωση. Η Κομισιόν εξετάζει λεπτομέρειε για το πώ θα απλοποιηθεί περαιτέρω η κινητικότητα προσώπων μεταξύ Ένωση και Τουρκία, ειδικά μέσω μια γρήγορη εφαρμογή του νέου κώδικα βίζα τη Ένωση, κάτι το οποίο θα έχει πρακτικέ βελτιώσει για όσου συζητούν βίζα από την Τουρκία. Επίσης η Κομισιόν ε, σκοπεύει να μπει σε έναν διάλογο ο οποίο θα οδηγήσει σε περισσότερη κινητικότητα μόλις μας δώσει το πράσινο φως το Συμβούλιο. Όμως ε, το να ολοκληρωθεί η σχετική συμφωνία με την Τουρκία νομίζω απαιτεί ένα, είναι ένα προαπαιτούμενο. Благодаря, господин председателстваш. Благодаря на всички колеги Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεχούχτ για τις εξαιρετικά θετικές ε, συστάσεις του και για τις χρήσιμες ε, θέσεις που έλαβε σε ό,τι αφορά την έκθεση της οποίας ε, έχω την τιμή να είμαι Η συζήτηση νομίζω οδηγεί στο συμπερισμό ότι οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας στο εμπορικό, στον εμπορικό και οικονομικό τομέα είναι θετικές για τις δύο πλευρές. Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη να εξελιχθούν ξεκάθαρα οι σχέσεις αυτές. Σκέφτομαι και κάποια ερωτήματα που έθεσαν ορισμένοι συνάδελφοι κατά πόσον οι σχέσεις αυτές συνδέονται ή όχι με την πιθανή προσχώρηση της Τουρκίας στην Ένωση. Η θέση μου είναι η εξής. Όσο πιο θετικά και επιτυχημένα προχωρούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο πιο επιτυχής θα είναι και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Βεβαίως και οι δύο πλευρές έχουν πολλή δουλειά ακόμα για να μπορέσουν να εφαρμόζονται οι ρήτρε που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως. Πιστεύω ωστόσο ότι πρέπει να έχουμε μια έντιμη και αντικειμενική στάση και από τις δύο πλευρές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι μετέσχουν στη συζήτηση. Έχω την άποψη ότι όλα τα προβλήματα που τέθηκαν στην σημερινή συζήτηση θα μελετηθούν προσεκτικά από την Επιτροπή και πιστεύω ότι χάρη στον ε, μηχανισμό διαβούλευσης Τελωνιακής Ένωσης όλα τα εκκρεμή προβλήματα θα ε, βρουν μία λύση σε πνεύμα καλής θέλησης για να επιληθούν ταχύ. Ευχαριστώ εκ νέου. Αύριο στις 12. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημερινή σε διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας ε, Ντελάνγκ, εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης